Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου, είναι μεγάλη εκπληξή μου που βρίσκομαι στην ε, έδρα του Πρόεδρου. Καλώς ήρθατε. Σας έχουμε διανύμει από 1η Ιουλίου την ημερησία διάταξη σε σχέδιο και όπως συμφώνησαν η επικεφαλής των Προέδρων Επιτροπών προτείνεται αναβολή της ψηφοφορίας για την έκθεση Τσασκόφσκι μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος δε συμφωνεί. Εγκρίνεται. Α, ο κ. Νταφ. Μα γιατί, γιατί αναβάλουμε την ψηφοφορία και ξανά και ξανά μάλιστα. μου είπαν ότι η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών επιθυμεί να συζητήσει το θέμα πριν να ψηφίσουμε. Ειλικρινώς όμως, Άντριου, δεν έχω καμία ειδική ενημέρωση. Και αν υπάρχει θέμα που πρέπει να συζητηθεί, θέστε το σας παρακαλώ υπόψη των συντονιστών αύριο. Ωραία λοιπόν, προχωρώ. Ο κύριος Μπροκ λόγω αεροπορικών κολλημάτων δεν θα μπορέσει να προσέλθει σήμερα. Δεν έχει λοιπόν νόημα να συζητήσουμε το υπαριθμό 6 της ημερησίας διατάξεως απουσία του εισηγητού. Καλύτερα να γίνει η σύντομη συζήτηση αύριο πριν από την ψηφοφορία όταν ο κύριος Μπρόκ θα μπορεί να προσέλθει κάπως νωρίτερα στη συνάντησή μας παρόλο που ταυτόχρονα διεξάγεται συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών ε, σας βρίσκει σε αυτή η αλλαγή. Δεν βλέπω κανέναν να ενίσταται, συνεχίζω λοιπόν. Οι καφέδες έχουν έρθει. Αύριο στο 11 διάφορα ο ίδιος ο κύριος Τρζασκόφσκι θα υποβάλει σχέδιο εκθέσεως για την διαθεσμική συμφωνία και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις ή άλλες επιθυμίες τροποποίησεων, θα θεωρήσω ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη με τις τροποποίησεις που σας ανακοίνωσα. Δεν βλέπω ενστάσεις. Συνεχίζω λοιπόν από την προηγούμενη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Συνταγματικών ενετάχθη η Κροατία και με μεγάλη χαρά υποδέχομαι δύο νέα μέλη της Επιτροπής μας, την κυρία Μπούσιτς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κυρία Πέτροβιτς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Καλώς ήρθατε στις δύο κυρίες. Θέμα 2, ανακοινώσεις του Προέδρου και πρώτα διαδικασίες κυρώσεως. Θα βρείτε το σχετικό πίνακα για το που βρίσκονται οι διαδικασίες κυρώσεων διαφόρων συνθήκων. Αυτά μόνον πληροφοριακός. Δεύτερο, διορισμός εισηγητών. Την προηγουμένη εβδομάδα έγινε γραπτή διαβούλευση μεταξύ των συντονιστών που έδειξε ότι εμφανίζεται συνένεση γύρω από την πρόταση του Λαϊκού Κόμματος σχετικά με τα της ε, συνθήκης που τα έχει δεχτεί και η διάσκεψη των Πρόεδρων. Προτείνω να εγκριθεί. Ωραία, δεν έχετε ούτε εδώ ενστάσεις. Θέμα υπαριθμών 3. Ο οργανισμός Ευρωπόλ. Η ε, κυρία Τέιν ορίστηκε τον Μάιο του 2013 ως εισηγήτρια γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Θεμελιδών Ελευθεριών για την νομοθετική αυτή πρόταση που προβλέπει νέο καθεστώς της Ευρωπόλ σύμφωνα με διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Η εμπλοκή της ΑΦΚΟ είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που διεξάγεται σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Τρία εθνικά κοινοβούλια του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ισπανίας ενέκριναν πρόσφατα ε, ψηφίσματα που λένε ότι δεν ε, συμβαδίζουν οι προτάσεις αυτές με το κοινοτικό κεκτημένο. Το ίδιο Σλοβενική και Πορτογαλική Βουλή που έχουν υποβάλει σχετικές προτάσεις. Αν θέλετε να εξετάσετε τα έγγραφα αυτά, να έρθετε σε επαφή με την γραμματεία. Τώρα, θα παρακαλέσω την κυρία Τέιν να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδοτήσεως και μετά θα ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές. Εάν κάποιος εξημών επιθυμεί να λάβει το λόγο, παρακαλώ να μας το γνωρίσει τώρα για να μπορέσω να μοιράσω το χρόνο. Κυρία Τέιν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Ευρωπόλ από το 2009 είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 2005 και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Με τον κανονισμό προτείνει η Κομισιόν συγχώνευση των δύο οργανισμών με σχετικά προγράμματα ανταλλαγής, εκπαιδεύσεως εθνικών υπαλλήλων, την μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπόλ ώστε αυτή να μπορεί να υποστηρίζει περισσότερο τις εθνικές αστυνομικές αρχές και καθεστώς προστασίας δεδομένων που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του εντεταλμένου την προστασία των, των, των προσωπικών δεδομένων. Άλλο σημαντικός στόχος της προτάσεως της Κομισιόν, με συγχωρείτε θα σας διακόψω, έχω έχω σχόλια από τους διερμηνείς που μου λένε ότι σας παρακαλούν να επιβραδύνετε το ρυθμό σας. Άλλος στόχος, όπως είπατε και εσείς, είναι η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπόλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούν στη βάση ετησίων εκθέσεων να ενημερώνονται. Εκτός αυτού προβλέπεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τα καθήκοντά του ως αρχή του προϋπολογισμού για το πολιετές πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπόλ και να ακροάτε των υποψηφίων για τον διορισμό στη θέση του Προέδρου της Ευρωπόλ. Την τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, είχαμε ήδη συζητήσει την πρόταση κανονισμού και οι συνάδελφοι εδώ της Επιτροπής Συνταγματικών τάχθηκαν κατά τη συγχώνευση των δύο οργανισμών. Έτσι λοιπόν εγώ στη γνωμοδότησή μου προβλέπω με τροπολογίες την ανατροπή αυτής της ιδέας της συγχωνεύσεως, δηλαδή οι δύο οργανισμοί να παραμείνουν ξεχωριστοί. Συμφωνήσαμε επίσης ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερη αξία στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών εδώ και μήνες ασχολείται με θέματα προστασίας δεδομένων. Για την προστασία δεδομένων λοιπόν εγώ έχω προβλέψει μια γενική απλώς τροπολογία διότι αλλιώς θα είναι πολύ ευρύ το κείμενο και θα μπαίνει και στα χωράφια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Κυρίως μιλούμε εδώ για τις διατάξεις περί λογοδοσίας απέναντι στο Ευρωπαϊκό αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια και μια πιο αποτελεσματική συνεργασία. Εγώ εξέτασα και πάλι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει και κάποιες ανεξάρτητες αρμοδιότητες. Αλλά αυτό φαίνεται πως δεν γίνεται, γιατί στην παράγραφο 88, στο άρθρο 88, παράγραφος 2, λέει ότι στον έλεγχο συμμετέχουν οι εθνικές βουλές. Από αυτό προκύπτει σαφώς ότι η λογοδοσία δεν μπορεί παρά να είναι από κοινού απέναντι στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβουλία. Το δε πρόβλημα στο παρελθόν ενέκειτο στο ότι στο παρελθόν τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν άσκησαν επαρκώς τον έλεγχο ή πάντως φάνηκε ότι ήταν δύσκολο. Έχω λοιπόν κάνει ορισμένες τροπολογίες για την υποχρέωση λογοδοσίας της Ευρωπόλ και δεν προβλέπω και κανένα νέο οργανισμό, διότι και αυτό ήταν εδώ η άποψη όλων, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τις, ενώ μάλλον δεν ε, πρότεινε νέα διαδικασία η εισηγητια διότι όλοι συμφώνησαν την προηγούμενη φορά ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες αυτά, ανα, ανακούσω τους συναδέλφους. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών μέχρι τις 5 Ενάτου. Η συζήτηση των τροπολογιών θα διεξαχθεί στις 15 Ενάτου και η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 15 Δεκάτου στην ΔΕ Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών τον Νοέμβρη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα μιλήσει κάποιος εξ αυτών. Α, θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γκυλιόμ πρώτα, γιατί ακόμα δεν βλέπω από το Λαϊκό Κόμμα. Ή μάλλον εσείς, και θέλετε να μιλήσετε εξ ονόματος των Πρασίνων, ωραία. Μετά λοιπόν από την κυρία Γκυλιόμ. Όχι, εσείς δεν θέλετε. Κυρία Άγνιου, εσείς. Ναι. Ωραία, μετά λοιπόν από τους άλλους που προανέφερα και μου μένει μόνο ο Άντζιου Νταφ, που θα δώσω, στον οποίο θα δώσω λόγο τελευταίο. Κύριε Γκυλιόμ, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μας είπε η κυρία Τάιν ε, ότι εργαζόταν εδώ και αρκετούς μήνες γι' αυτό και για να εξετάσουμε αύριο την έκθεση των Άλλωστε το είχα πει επειδή 17 Ιουνίου δεν ήμουν εγώ εκεί όταν ξεκίνησε η συζήτηση στην ΑΦΚΟ για αυτή την πρόταση για τη συγχώνευση της υπόλοιπης Europol και η ομάδα μου είπε ότι είναι σταθερά κατά αυτής της πρότασης και νομίζω κύριε μου ότι το ίδιο φρονείτε και εσείς και ότι κάποιες από τις απολογίες προς τα αυτά κατεύθυνση πηγαίνουν όπως είπαν και τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Λίμπε και άλλων κατά τη συγχώνευσης αυτών των δύο. Αυτό λοιπόν. Κάτι ακόμα που θέλω να πω. Η ΑΦΚΟ θα πρέπει να συγκεντρώσει προσπάθειά τη για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, των δραστηριοτήτων τη Europol και να υπάρχει ένα σχέδιο εργασία τη Europol ε, και να υπάρξει μια συνάντηση με το Ευρωκοινοβούλιο, κάποιε παρόμοιε προτάσει. Ε, και για τους τρόπους, για τις προτάσεις, πώς θα γίνουν αυτά, νομίζω ότι τα αντιμετωπίζετε κατάλληλα μέσω διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και πώς τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν να παίξουν ε, σημαντικότερο ρόλο στις όλες εργασίες. Για να προχωρήσουμε δε γρήγορα στην έκθεση αυτή, να πούμε ότι υποστηρίζουμε αυτές τις προτάσεις ε, στην ομοδοτησή σας ε, για τον έλεγχο τον μεγαλύτερο, τον κοινοβουλευτικό, τον ευρύτερο. να γίνεται συνήθως και για την κατάρριξη προτάσεων που έχει να κάνει με συγχώνευση σε Πολ και Europol και ε, λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον ε, Ευρωπαϊκό Ελεγκτή Δεδομένων όπως αναφέρεται στην εκθεσή σας και σημαντικό είναι να το δούμε κάτω από το, αυτό το πρίσμα λοιπόν θετικό μάλλον για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κυρία μου. Γκέραλτ από τους πράσινους, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι και εσείς κυρία Τάιν. Σημαντική αύξηση ποινικών αδικημάτων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στην κύβερνο εγκληματικότητα πλήσιμο χρημάτων και ούτω καθεξής τα τελευταία δέκα χρόνια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η εργασία της Ευρωπόλ, όπως και των Εθνικών Αστυνομικών Αρχών, να εξεταστεί από εμά ιδίως ό,τι αφορά την αποδοτικότητά της. Επίσης να εντοπιστούν τομείς συνεργασίας και μαζί με την Τσίπολ που παίζει κέριο ρόλο. Ωστόσο, Είμαι επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση της συγχωνεύσεως για ένα αριθμό λόγων που ήδη αναπτύχθηκαν από την κυρία Τάιν. Εξ ονόματος της ομάδος μου έχω να πω ότι αυτή η βραχύτατη σύνοψη που έκανε η κυρία Τάιν, αλλά οι προτάσεις της είναι αρκετά ανεπτυγμένες στο σχέδιό της, μας βρίσκουν σύμφωνους και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο. Πολύ καλά. Εσείς δεν θα πάρετε λόγο, κύριε Σμιθέτη, δεν είναι. Ο κύριος Άκη, Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλώντας για την ενίσχυση της Europol, η οποία για πολλούς από εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά προβληματική οργάνωση. Αυτό που με προβληματίζει στην πρόταση αυτή είναι μία συγκεκριμένη πρόταση. Εγγυάται ότι ο επέπτυξης προσωπικών δεδομένων της Ευρωπόλ έχει πλήρη ανεξαρτησία, μπορεί να δράσει αποτελεσματικά και έχει επαρκείς εξουσίες ή αρμοδιότητες παρέμβασης. Δεν μου αρέσει αυτή η πρόταση. Μπορεί να παρέμβει για να πάρει στοιχεία από το DV Λέει ή από το, τα τελωνία και την εφορία της αυτού μεγαλειότητος ή από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να επιτρέψουμε σε ένα άτομο να έχει πρόσβαση σε τέτοιου πληροφορίες. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό κατά τη γνώμη μου. δεν υπάρχει αστυνομικός φορέας όπου να μην υπάρχει τουλάχιστον ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και θέλω όλα, όλα αυτά τα στοιχεία να παραμένουν εντός της επικράτειας της χώρας μου και να μην ταξιδεύουν αλλού. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Άντριου Νταφ. Ε, όμως, το ΕΛΚ δεν έχει συμβάλει στο σημείο 3. Αν κάποιος από το ΕΛΚ θέλει να συμβάλει, να μου το πει λίγαν συντόμως, αλλιώς μόλις μιλήσει ο Άντριου θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Άντριου, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να δούμε, ή τουλάχιστον θα ήθελα εγώ να δω, τις τρεις αιτιολογημένες ε, γνωμοδοτήσεις από τα ε, τμήματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, στα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Μπορείτε να τα ε, μοιράσετε στα μέλη της Επιτροπής ή τουλάχιστον να μου δώσετε εμένα ένα αντίγραφο. Ε, είναι περίεργο το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος κανονισμός ο οποίος να παραβαίνει υποτίθεται την αρχή της επικουρικότητας όταν ακριβώς τίθεται θέμα, το, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι τα διασυνοριακά αστυνομικά ζητήματα. Περίεργο λοιπόν τα λέγεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει με ενδιαφέρει να δω τις εκθέσεις αυτές τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να μας επαναλάβει τα επιχειρήματα. Γιατί πιστεύουμε, γιατί φρονούμε ότι αυτά τα δύο όργανα, αυτοί οι δύο φορείς δεν θα πρέπει να συγχωνευτούν. Η τεκμηρίωση της Επιτροπής πίσω από την πρότασή της για τη συγχώνευση αυτών των δύο φορέων είναι η εξής. Είναι μια τεκμηρίωση μάλλον που φαίνεται αρκετά εύλογη, λογική, δίκαια. Πράγματι, ε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχουμε ε, σχέση κόστους ωφέλειας πολύ καλύτερη μετά από τη συγχώνευση αυτών των δύο οργανισμών. Δεν βλέπω γιατί η ε, κατάρτιση και η εκπαίδευση της αστυνομίας, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος, γιατί η ξεχωριστή κατάρτιση ε, και εκπαίδευση είναι εγγενώς ε, κάτι το κακό. Καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούμε. Να ξαναδούμε τα ουσιαστικά επιχειρήματα που έχουμε για να αντιταχθεί κανείς στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτον, ως προς την τροπολογία 16. Είμαι κάπως προβληματισμένος, διότι στην παράγραφο 2α, στην τρίτη παράγραφο δηλαδή αυτής ε, της τροπολογίας, λέτε αρχικά ότι ο έλεγχος θα ασκείται γράφεται exerted, αλλά μάλλον εννοείται asserted, θα επιβεβαιώνεται δηλαδή ο έλεγχος από ένα κοινοβουλευτικό όργανο. Και στο τέλος λέτε ότι τον έλεγχο θα το οργανώνει ε, η υφιστάμενη κοινοβουλευτική δομή. Υπάρχει εκεί δηλαδή μια κάποια αμφισημία. Ε, γιατί ακριβώς πράγμα μιλούμε. Εάν θεωρήσουμε ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει ήδη επιτύχει σε μεγάλο βαθμό ε, την διακοινοβουλευτική συνεργασία με ε, τις ομόλογες επιτροπές της στα Εθνικά Κοινοβούλια, Και αν θεωρούμε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επισημοποιήσουμε αυτή την πρακτική, τότε έχει καλός δεν θα έπρεπε τότε να μιλούμε ότι τον έλεγχο θα τον επιβεβαιώνει, θα τον επικυρώνει ένα διακοινοβουλευτικό ε, σώμα, γιατί αυτό υπονοεί τη δημιουργία ενός ε, καινούριου φορέα. Ε, ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσετε τη διατύπωση. Ευχαριστώ. Ο, ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Χέφνερ, είπατε ότι θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Κυρία Χέφνερ. Συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρος. Ο κ. τελικά μετά από την ε, σύντομη διακοπή. Έρχομαι σε δύο θέματα που ανέφερε ο Άντριο Νταφ και ίσως μάλιστα να επεκταθώ και λίγο περισσότερο. Δεν είναι σύνηθες οι εθνικές βουλές να προβάλλουν απέναντί μας ένσταση επικουρικότητας και να κάνουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που εκφράζουν την άποψη ότι κάτι, κάποιο, κάποια νομοθετική πράξη που εγκρίνεται εδώ υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η συνθήκη και διεισδύει στις νομοθετικές αρμοδιότητες των χωρών μελών. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να γνωρίζουμε τις γνωμοδοτήσεις που υποβάλλουν οι Εθνικές Βουλές και να τις περιλαμβάνουμε, να τις μελετούμε και να τις περιλαμβάνουμε στο σκεπτικό μας. Αυτό μάλιστα όχι μόνο στην περίπτωση την οποία ανέφερε ήδη ο κ. Ντάφαλα και τακτικά στο μέλλον στα πλαίσια της ορθής έντιμης ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τέτοια έγγραφα από εθνικά κοινοβούλια, να μας υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά έγγραφα, ώστε να μπορούμε και να τα εξετάσουμε και να αναφερθούμε, να παραπέμψουμε σε αυτά. Ένα άλλο σχόλιο, πιο γενικό, έρχομαι στην τροπολογία υπαριθμών 8 που λέει ότι ο κοινός κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της Ευρωπόλ θα γίνεται μέσα στα πλαίσια των διακοινοβουλευτικών δομών. Εδώ επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι αυτές οι φυστάμενες διακοινοβουλευτικές δομές ως δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος δεν είναι ούτε ευτυχείς ούτε αποδοτικές. Σας προσκαλώ λοιπόν να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο αποτελεσματικές κοινέ διαδικασίες ελέγχου όπου θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Θα είναι πράγματι χρήσιμο οι αιτιολογημένες γνώμες να περιλαμβάνονται στα έγγραφα που λαμβάνουν τα μέλη της Επιτροπής. Μόλις μίλησα με τον γραμματέα, ο οποίος συμφώνησε. Τώρα ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ. Από αυτά που είπατε αρχικά, είχα κατανοήσει ότι θέλετε να μην μιλήσει παραπάνω από ένας βουλευτής από κάθε πολιτική ομάδα. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει περισσότερος, ε, ε, περισσότερο περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο. Και έτσι λοιπόν, ε, έστω και μίλησε πριν ο κύριος Άγνιου, λαμβάνω το λόγο και εγώ. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, η Ευρωπόλ βασίζεται στη συμφωνία πλαίσιο παλαιότερης συνθήκης και τώρα πάει να γίνει κανονισμός. Αυτό αλλάζει τη νομική βάση, τη νομική θεμελίωση μέσα στην συνθήκη και επηρεάζει την χώρα μου, την Δανία που έχει opt-out που δεν θα έχει εφόσον είναι κανονισμός. Και άλλες χώρες το ίδιο. Πώς, ε, μπορείτε να πείτε κάτι για το πώς θα ληφθεί αυτό υπόψη στη νέα πρόταση. Πώς θα επηρεάσει μια χώρα η οποία διαθέτει εξαίρεση, opt-out, όταν θα αλλάξει ε, η νομική βάση της Ευρωπόλ. Μάλιστα. Κυρία Τάιν, θέλετε να απαντήσετε στις διάφορες παρεμβάσεις. Ε, ναι, ευχαριστώ βεβαίως. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ για την ε, λίγο πολύ συμφωνία από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα έρθω τώρα με τη σειρά στις ε, διάφορες παρεμβάσεις. Ο κύριος της ECR είπε ότι είναι θεμελιωδώς αντίθετος σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων κτλ. Νομίζω ότι πρόκειται για θεμελιωδώς άλλη πολιτική άποψη από αυτή που έχω και εγώ ως φιλελεύθερη και παρακολουθώντας την συζήτηση τελευταία από τις διάφορες κατασκοπικές δραστηριότητες και από τις ΗΠΑ αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο σε βάρος άλλων χωρών. Τότε και εγώ ως Γερμανίδα ε, δηλώνω ότι έχω μια πολύ διαφορετική πολιτική αντίληψη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εντεταλμένος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτός να είναι απόλυτα ανεξάρτητος και να έχει ευρύτατες αρμοδιότητες. Νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διάστασης απόψεων μεταξύ διαφορών πολιτικών σχηματισμών. Βλέπουν τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά, ιδίως σε ό,τι αφορά την αστυνομική συνεργασία. Όμως, η αντιδράση των πολιτών, ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον στην πλειονότητα των χωρών μελών, δείχνει, δείχνουν μάλλον οι αντιδράσεις, ότι οι πολίτες αποδίδουν ιδιαίτερη αξία σε μια εκτεταμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και όλη αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων κάπου τους έχει φανεί καθαρά υπερβολική. Δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε γιατί ξεκινάμε από διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Όσον αφορά την πρόταση της συγχωνεύσεως, σύνδεξη λέει εδώ στα γερμανικά, ε, το βασικό επιχείρημα είναι ότι θα εξοικονομηθούν χρήματα. Αυτό το αμφισβητούν ορισμένοι ότι θα προκύψουν κάποιες εξοικονομήσεις. Ούτως ή άλλως και εμένα δεν μου αρέσουν πολύ οι πολυπληθείς οργανισμοί, που έχουμε και θεωρώ ότι πρέπει κάπως να επιτηρούνται, να εποπτεύονται. Αλλά η αστυνομική δραστηριότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι διαφορετικός τομέας και άλλο η εκπαίδευση, άλλο η καθαρά αστυνομική δραστηριότητα και σε πολλέ χώρε μέλη είναι ξεχωριστέ. Οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε και την προηγούμενη φορά τάχθηκαν κατά και για την ομάδα και μάλλον για την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπω είπα, εκφράζει ομόφωνα τη γνώμη αυτή. Γι' αυτό και πρότεινα αυτά που πρότεινα ως απηχούντα την άποψη της πλειοψηφίας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Βουλών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν δηλαδή τώρα θα θεωρηθεί ως ένα ενίο σώμα ή όχι, εγώ κάθισα και προβληματίστηκα πολύ. Για παράδειγμα, πόσο συχνά πρέπει να συνέρχονται τα όργανα αυτά. Αλλά μου είπαν οι σύμβουλοι ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν έχουμε το δικαίωμα μέσα σε κανονισμό να επιβάλλουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια να έρχονται τόσες φορές το χρόνο εδώ. Έχουμε τη συνεργασία αυτή με τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι και πολύ δύσκολη και εξαρτάται για παράδειγμα και αν, από το αν υπάρχει επαρκώ επαρκώς μεγάλη αίθουσα και γι' αυτό δεν συναντώμεθα και τόσο συχνά με τα Εθνικά Κοινοβούλια διότι υπάρχει και πρόβλημα χώρου και πρόβλημα χρόνου. Και βεβαίω και από θεσμική άποψη δεν επιτρέπεται να βάλουμε τέτοιο περιεχόμενο σε ένα κανονισμό. Αλλιώς εγώ πολύ ευχαρίστως θα έγραφα εδώ ότι θα πρέπει να συναντώμεθα αναδίμηνο. Όμως και η Κομισιόν και το Συμβουλίο μου είπαν «Α, όχι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται». Εγώ λοιπόν ψάχνω να βρω μια ενδιάμεση λύση όπου θα μπορεί η συνεργασία να ενταθεί Προσπάθεια, λοιπόν χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη στα γερμανικά γκρέμι που μεταφράζεται στα ελληνικά ως όργανο να δείξω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο επίπεδο όπου να συναντώνται τα, τα κοινοβουλία. Αυτό θεωρητικά μπορεί να γίνει. Τώρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι αφενός δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αφετέρου βέβαια θα είναι καλό να συναντώμεθα περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα της επικουρικότητας, στην ε, νομική μας επιτροπή μας υποβάλλεται πάντοτε αυτομάτως οποιαδήποτε ένσταση επικουρικότητας. Βέβαια, εμεί είμαστε και πολύ πιο αρμόδιοι για τον έλεγχο τη επικουρικότητας, αλλά μπορεί ίσως να γίνει το ίδιο και εδώ. Εγώ τάσομαι πάντω υπέρ. Το άλλο είναι ότι στη Γερμανία ήδη έχουμε το πρόβλημα ότι ολόκληρη η αστυνομική, υπόθεση αστυνομικής εργασίας είναι καθαρά θέμα των κρατηδίων, των ομόσπονδων χωρών μας δηλαδή. Αυτή η συνεργασία της Ευρωπόλ θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη Γερμανία. Ο κανονισμός και όπως είναι, διότι ορισμένα καθήκοντα κρατηδίων δεν θα μπορούν να, να συνεχίσουν να ασκούνται όπως μέχρι τώρα. Και γι' αυτό προέκυψε και για μας αυτή η ένσταση ή μομφή επικορικότητας. Για μας είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και συνταγματικότητας. Τέλος πάντων η ένσταση αυτή ήρθε, η μομφή δηλαδή. Μια φορά πάντως εμείς με την νομική επιτροπή πήγαμε στην ίδια τη Χάγη και εξετάσαμε τις υποθέσεις της Ευρωπόλ. Διεξάγονται για παράδειγμα έρευνες ταυτόχρονα μέσα στην ίδια μέρα σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη από πολύ στενή συνεργασία. Άρα, εφόσον ε, δραστηριοποιείται η Ευρωπόλ, αφαιρούνται και αρμοδιότητες από άλλες αστυνομικέ αρχές. Αυτό ε, έχει τον κίνδυνο να μπουν πολύ στα χωράφια συνταγματικών αρμοδιοτήτων των χωρών μελών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ε, ωραία, ευχαριστώ πολύ κυρία Τάιν. Καλώς. Πρέπει τώρα να υιοθετήσουμε το χρονοδιάγραμμα για τη γνωμοδότηση αυτή θα σας προτείνω τα εξή γιατί έχω δει και το χρονοδιάγραμμα της ε, Βασικής Επιτροπής. Υποβολή τροπολογιών 5 Σεπτεμβρίου στις 12. Ε, εξέταση των τροπολογιών 16-17 και ψηφοφορία 18 Οκτωβρίου. Συμφωνείτε? Τότε θεωρώ ότι έχουμε συμφωνήσει. Σας ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε. Στο σημείο 4 της εμερήσιας διάταξης Γενικός Προπολογισμός του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική χρήση ε, του 2012 με εισηγητή τον κύριο Messerschmidt. Έχουμε υιοθετήσει ήδη γνωμοδότηση που έχει συντάξει ο κύριος Σμιτ. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει ε, γνωμοδότηση αλλά και τροπολογίες στο σχέδιο προϋπολογισμού. Στη, στη σημερινή συνεδρίαση ο εισηγητής έχει ε, προετοιμάσει ένα σχέδιο διατάξεων γνωμοδότησης και έχουμε κάποιες βασικές προκαταρτικές τροπολογίες που βασίζονται στα στοιχεία του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό το κύριο Μέσο Σμιτ λοιπόν να παρουσιάσει τις προτάσεις του καταρχάς και αν θέλουν και τα υπόλοιπα μέλη να συμβάλλουν να μου το ε, καταστήσουν σαφές. Κύριε Μέσο Σμιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε πριν από ένα μήνα υιοθετήσαμε τη γνωμοδότηση ως προς την απόφαση της ΑΦΚΟ για την Οικονομική χρήση 2014. Μετά την έγκριση της γνωμοδότησης, αυτήν την μετέτρεψα σε τέσσερις τροπολογίες που θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει και να σας έχουν μοιραστεί ή κάτι το οποίο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων λογαριασμών χωρίς να αυξάνει, να επηρεάζει κατά τη το προϋπολογισμό. Πρώτον, η τροπολογία μας έχει να κάνει με την ενημερώση των πολιτών για ε, την έλευση των εκλογών προκειμένου να υπάρξει περισσότερη προσέλευση κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών του χρόνου. Δεύτερον, που είναι βασικά το ίδιο. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί του χρόνου για το τι θα έχει γίνει. Και αυτό έχει τροποποιηθεί, έχει προσθεθεί δηλαδή ως τροποποίηση στη γενικότερη πρόταση και το ίδιο ισχύει και με την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις δραστηριότητες του 2013, αλλά εκτείνεται και σε ένα πιο ευρύ πεδίο ε, προσπαθώ εδώ να υλοποιήσω αυτό που πρότεινε ο κύριος Χέφνερ για να ξέρουμε ακριβώς πώς έχει δουλέψει αυτό το πράγμα, ποια ήταν τα εμπόδια, ε, πώς μπορούν να αρθούν και να επιληθούν τα προβλήματα. Κάτι το οποίο ε, θα οθήσει αυτή την πρωτοβουλία ακόμη υψηλότερα στο μέλλον. Αυτές λοιπόν είναι οι υποδείξεις και οι προτάσεις. Ευχαριστώ θερμά τη Γραμματεία για τη βοήθειά της. Εάν θέλει κάποιος και άλλες τροπολογίες να υποβληθούν, αφού λείπει και η πρόταση του Συμβουλίου, έχουμε χρόνο πιστεύω έναν κάποιο χρόνο, οι υποδείξεις σας είναι ευπρόσδεκτες. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κανείς δεν ζήτησε τον λόγο. Ε, όση ώρα μιλούσατε κύριε Μέσο Σμίτ, αυτό μάλλον δείχνει ότι συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Συγχαρητήρια. Ε, κοιτάζω και βλέπω ικανοποιημένα πρόσωπα στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. χρονοδιάγραμμα, η υιοθέτηση της γνωμοδότησης. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια σύντομη συνεδρίαση Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου από τη 1 έως μια και μισή, μια έκτακτη συνεδρίαση για να το εγκρίνουμε αυτό, ε, προτινόμενη ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών και για τα δύο είναι η Τετάρτη 24 Ιουλίου ε, στα, το μεσημέρι. Ε, τις παραμονές δηλαδή των διακοπών. Έχετε σχόλια για το χρονοδιάγραμμα. Εάν όχι, θεωρώ ότι υπάρχει συμφωνία. Καλώς. Ευχαριστώ. So, Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση έκθεση για τις έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμάστε ότι η έκθεση αυτή ότι η έκθεση αυτή συζητήθηκε στη συνεδρίασή μας στις 8 Ιουνίου. 124 τροπολογίες υποβλήθηκαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Δεν έχουμε μετάφραση των τροπολογιών αυτών στις υπόλοιπες γλώσσες. ως συνεισηγητής κατάλαβα τις αγγλικές τροπολογίες και τις γαλλικές, αλλά όχι τις γερμανικές και τις υπόλοιπες. Ο κύριος Χέφνερ που είναι επίσης συνεισηγητής με βοήθησε για τις γερμανικές. Ελπίζω όλοι να έχετε μπορέσει να καταλάβετε τις ε, τροπολογίες. Να ξεκινήσω εγώ κύριε Χέφνερ ως πρώτος συνεισηγητής και εσείς μετά για να συνοψίσετε. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το τμήμα της διαδικασίας μόνο και μόνο για να ακούσουμε τη συνεισφορά που έχετε να κάνετε εσείς, τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε υποβάλει πολλές τροπολογίες, κάποιες είναι χρήσιμες και κάποιες δεν βοηθούν καθόλου και το λέω αυτό απολύτως, με απόλυτη ειλικρίνεια κάποιες τροπολογίες άσκησαν κριτική στους αριθμούς, στα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε εμείς, εγώ και ο Γκέρελτ, στην έκθεσή μας. Αριθμητικά στοιχεία, νούμερα που αποτιμούν το κόστος του να υπάρχει έδρα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και θα έλεγα ότι όσοι ασκούν κριτική ε, στα στοιχεία που χρησιμοποιούμε, τείνουν να είναι τα ίδια μέλη που εμπόδισαν το Κοινοβούλιο να έχει ακριβή αριθμητικά στοιχεία στο παρελθόν. Συμφωνούμε απολύτως. Απουσιάζουν πληροφορίες ακριβείς για τη διατήρηση των δύο εδρών. Γιατί? Διότι δεν θέλουν να διατεθούν αυτά τα νούμερα δύο βασικές ομάδες στο Κοινοβούλιο. Μόνο πέρσι υπήρξε ευρεία συνένεση ε, μεταξύ των απλών βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου ότι ε, χρειάζεται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο από πλευρά κυρίου Χέφνερ που αποτελεί και τη βάση των αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων μας και κάποιες από τις τροπολογίες που υποβάλλατε εσείς, τα μέλη, ε, ζητούν περαιτέρω διερεύνηση για το κόστος ύπαρξη δύο κτηρίων και χαίρομαι για αυτές τις τροπολογίες πραγματικά. Θέλω όμω να πω και το εξή. Δική μα θέση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία έδρα και να αποφασίσει το Κοινοβούλιο πού να είναι αυτή η έδρα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι θέλουμε μία έδρα στις Βρυξέλλες, ούτε λέμε ότι θέλουμε μία έδρα στο Στρασβούργο. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι βοηθητικό να έχουμε τροπολογίες που ζητούν να εκτιμηθεί το κόστος μόνο εάν μετακινηθεί η έδρα στο, στις Βρυξέλλες αν είναι να ερευνήσουμε, θα πρέπει να ερευνήσουμε και τα δύο. Ποιο θα ήταν το κόστος ύπαρξης μίας έδρας στις Βρυξέλλες μόνο και από την άλλη ποιο θα ήταν το κόστος ύπαρξης μίας έδρας στο Στρασβούργο μόνο. Και άργα θα είμαι ειλικρινή. Δεν είναι σκοπός της έκθεσης μας να πούμε πού θα πρέπει πραγματικά να είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έρχομαι τώρα στους κοιόδης εισηγητές η κυρία Λεγκρίπ ε, ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να συμβάλλει ε, στη συζήτηση σήμερα. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Εσείς. Κοιτάξτε. Θα ήθελα να μιλήσω, αλλά να μην εκπροσωπήσω την πολιτική μου ομάδα. Η απόψη μου είναι καθαρά προσωπική για το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσω ως εκπρόσωπος της πολιτικής ομάδας. Ο κύριος Δρούτσας. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Να σας πω ότι πράγματι μιλώ εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών ε, της σκιώδους εισηγήτριας. Είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα αυτό, ειδικότερα για ορισμένους συναδέλφους. Είναι προφανές ότι πολλές ιδέες και προσεγγίσεις υπήρξαν, πολλές και διαφορετικές από πολλούς συναδέλφους στη δική μου πολιτική ομάδα και τις σέβομαι όλες πλήρως. Να ξεκινήσω καταρχάς ευχαριστώντας τους δύο συνεισηγητές, τους κοιόδες εισηγητές, όλους τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες. Πρέπει να εκφράσω την έκπληξή μου για τον υπερβολικά υψηλό αριθμό τροπολογιών σε μία έκθεση η οποία έχει μεγάλη πολιτική αξία και έντονο συμβολισμό. Ε, έτσι έχει το πράγμα, όπως και να το κάνουμε. Προσωπικά θα προσπαθήσω να περιοριστώ μόνο στις ε, τροπολογίες που έχουν να κάνουν με θέματα αρχής. Έχω υποβάλει μόνο δύο τροπολογίες και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Μία που ε, θεσπίζει μία νέα αιτιολογική σκέψη η οποία αναφέρεται σε αυτό το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό, δηλαδή στον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό σε κάποιες ή πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία ε, επίσης η αιτιολογική σκέψη έχει να κάνει με το πόσο υπονομεύεται η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πόσο μάλλον που θα έχουμε ευρωεκλογέ ε, την επόμενη χρονιά. Σε λιγότερο από 12 μήνε. πρέπει να βάλουμε τα καλά μα για να κάνουμε τη βέλτιστη δυνατή εντύπωση στον Ευρωπαίο πολίτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει το παν για να φανεί όσο δυνατόν πιο αξιόπιστο στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη. Και αυτό είναι και το πνεύμα τη τροπολογία μου για την σύνταξη μιας νέα αιτιολογικής σκέψη. Η δεύτερη τροπολογία που υποβάλλω έχει να κάνει με κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, στην τελευταία μας συνεδρίαση, όταν εξετάσαμε την έκθεση αυτή. Είναι κάτι που είπα και από την πρώτη στιγμή, άλλωστε. Είναι κάτι που είναι και εξαιρετικά σημαντικό για εμένα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η συζήτηση και η εξέταση εναλλακτικών λύσεων για την αξιοποίηση των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν τελικά προκύψει μία μόνο έδρα, όπου και να είναι στο μέλλον, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κτίρια. Να το έχουμε εξετάσει. Τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη που ε, θα κληθούν να παρετηθούν από τη, μία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πράγματα που θα πρέπει να έχουμε εξετάσει εκ των προτέρων για να υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέω με πάσα ειλικρίνεια και εκφράζω την προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι και η πλειονότητα τη πολιτική μου ομάδα συμφωνεί, ενστερνίζεται την άποψη αυτή δεν θα είμαστε πολύ θετικοί έναντι των τροπολογιών που προσπαθούν να απορρίψουν τη γενικότερη προσέγγιση της έκθεσης ε, της τοποθέτησης επί της αρχής της έκθεσης αυτής, όπως το τονίσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση και να εμείνουμε σε αυτή. Δηλαδή, να μην μιλούμε για το ποια θα πρέπει να είναι η πόλη της μίας και μόνης έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο δικαίωμα αυτοοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αυτή είναι μια νέα προσέγγιση και θεωρούμε ότι είναι πιο χρήσιμη ε, για ε, την επίλυση του ζητήματος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, τροπολογίες από συναδέλφους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για την έκθεση αυτή είναι ευπρόσδεκτες και αυτές που τονίζουν την ιστορική και συμβολική αξία της πόλης του Σταυρασβούργου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αξιόλογες τροπολογίες και θα πρέπει να προσθεθούν στην έκθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνουν την ε, τοποθέτηση επί της αρχής που παρουσιάζει η έκθεση αυτή. Αυτά λοιπόν έχω να πω για τις τροπολογίες από πλευράς της πολιτικής μου ομάδας. Ε, με εκπλήσει κύριε Πρόεδρε σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μετάφραση όλων των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε κάποιες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι όλες. Παρακαλώ να το διαβάσετε στη γραμματεία, ώστε να μεριμνήσει να έχουμε τις μεταφράσεις όλων των τροπολογιών σε όλες τις, χώρες, σε όλες τις γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κύριε Νταφ, δεν βλέπω τον συνάδελφό σα κύριο Βίλτσεφ. Ίσως θα μιλήσετε εσείς εξ ονόματος των φιλελεύθερων. Δεν ξέρω, ας δούμε τι θα πω πρώτα. Και μετά θα αποφασίσουμε απαντά Για το θέμα της έδρας του Κοινοβουλίου. Δεν έχω ξαναλάβει το λόγο για αυτό το θέμα. Το μόνο που πιστεύω είναι ότι αυτή η υπόθεση του κόστους ίσως είναι υπερβολική. Εμένα με ανισχύει λιγότερο αυτό. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι η νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου. Και για να γίνουμε ένα πλήρες νομιμοποιούμενο κοινοβούλιο που ασκεί πλήρως τις εξουσίες του που προβλέπει η συνθήκη, χρειάζεται φυσική εγκύτητα με τα άλλα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο. Βρίσκονται απαραίτητα αυτά. Και έτσι όπως είμαστε κατακαιρματισμένοι σε δύο και αν βάλουμε και το Λουξεμβούργο τρεις πόλεις, αυτό το γεγονός και μόνο αποδυναμώνει το Κοινοβούλιο. Αυτό με ανισχύει πρωταρχικά. Τίθεται και το ερώτημα, εάν το Κοινοβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσει περί της έδρας του. Ο κύριος Δρούτσας το είπε αυτοοργάνωση. Δεν είμαι και βέβαιος ότι το έχουμε το δικαίωμα αυτό. Δεν βλέπω και κανένα θεσμικό προηγούμενο όπου κοινοβούλια να έχουν αποφασίσει από μόνα τους ποια είναι η έδρα των εργασιών τους. Εξάλλου με απασχολεί και η αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, που είναι αρχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και που μας δεσμεύει και που λέει ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με Συμβούλιο και Κομισιόν. Επίσης ανησυχώ σχετικά με το ότι υπό τις παρούσες συνταγματικές περιστάσεις Κοινοβουλίου και Ένωσης γενικότερα, τα δύο τμήματα της νομοθετικής αρχής θα πρέπει να γίνουν πιο ίσα, πιο ισότιμα. Δηλαδή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Για τους λόγους αυτούς, συμπεραίνω ότι αντιθέτως από την προσέγγιση των δύο εισηγητών, δεν έχουμε και ούτε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε ή ότι διαθέτουμε αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσουμε που συνερχόμεθα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να συναποφασίζουμε για το θέμα αυτό με το Συμβούλιο. Αυτό λέω και στην τροπολογία μου με τον αριθμό 90. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, γνωρίζετε όλοι ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη. Οφείλουμε να το δεχθούμε. Και εξεπλάγει που είδα στο σχέδιο εκθέσεως των δύο εισηγητών να δω τι κάνουν ακριβώς. Στην παράγραφο 2. Δεσμεύονται να αρχίσουν ή να προκαλέσουν αλλαγή της συνθήκης ενώ έχουμε το δικαίωμα να την εκκινήσουμε. Στην τροπολογία με 104 διατυπώνω σαφώς την αλλαγή που πρέπει να επέλθει στο οικείο άρθρο της συνθήκης που θεωρώ ότι είναι και ευκταία και αναγκαία αλλαγή. Όσοι θα γνωρίζετε υπάρχουν και άλλες εκθέσεις που κυκλοφορούν μέσα στο Κοινοβούλιο επί του παρόντος και που ζητούν αλλαγές στη συνθήκη. Θα πρέπει να φανεί η ΑΦΚΟ αρκετά τολμηρή και να περιλάβει μια ρητή πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαδικασία λήψη αποφάσεω για την έδρα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Άντριο, να σας απαντήσω για την πρόταση συνταγματικής αλλαγής ευθύς αμέσως. Θα θυμάστε ότι όταν οι συντονιστές συζήτησαν την έκθεση, εμείς θέλαμε αρχικά έκθεση που να προτείνει αλλαγή στη συνθήκη, ή διάσκεψη των Προέδρων το ανέτρεψε αυτό και είπε ότι μπορούμε να κάνουμε έκθεση ίδια Αν η ερμηνεία σα είναι σωστή, τότε δεν έχουμε ούτε καν αυτήν. Και γι' αυτό ο Γκέραρτ και εγώ δεν προτείνουμε συνταγματική αναθεώρηση ή αναθεώρηση της συνθήκης δηλαδή, αλλά προτείνουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση μα για να ανοίξουμε το δρόμο για την επόμενη έκθεση το 2014, εφόσον βεβαίω εγκριθεί. Θε να απαντήσει, Άντριου, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να συγκεντρωθούν τα πνεύματα της διάσκεψης των προέδρων των ομάδων, αν δουν επιτέλους πάνω σε χαρτί τι ακριβώς θέλουμε. Σύμφωνοι, λέει ο Πρόεδρος. Όσοι ήρθαν στις 4 η ώρα για την έκθεση αυτή, θα σας πω ότι αρχίσαμε λίγο νωρίτερα. Έχω μόνο τον κύριο Ράνζελ. Εσείς που είστε της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς, πώς θέλετε να μιλήσετε και Σόλτς, εσείς και μετά έχω τους άλλους, Σέφριν και λοιπά και ο Σάφνερ στο τέλος. Ράνζελ. Θα είμαι Είμαι λίγο απογοητευμένος με τις τροπολογίες που όχι μόνο αμφισβητούν κάποιες στατιστικές αλλά μάλιστα υποβάλλουν και εναλλακτικές στατιστικές που και αυτόν η μεθοδολογία είναι αμφισβητήσιμη. Εάν η βασική θέση είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε στατιστικές, Μιλώ τώρα από την οπτική γωνιά αυτών των συναδέλφων. Άμα λένε ότι δεν πρέπει να μιλούμε για στατιστικές, τότε γιατί υποβάλλουν εναλλακτικές στατιστικές. Τέλος πάντων, δεύτερο. Αν καταλαβαίνω καλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ, ίσως είναι μια τακτική διαφορά περισσότερο, μεταξύ ορισμένων που πιστεύουν ότι πρέπει να δούμε το θέμα αυτό ως ζήτημα υπαγόμενο στην συναπόφαση ή ως ζήτημα προνομίου ή εξουσίας του Κοινοβουλίου. Φαίνεται να υπάρχουν αυτές οι δύο διστάμενες απόψεις. Και πάλι εγώ τονίζω ότι εγώ δεν νομίζω ότι η συναπόφαση είναι καλή περίπτωση εδώ, για δύο λόγους. Διότι αν δεχθούμε, αν δεχθούμε ότι δεν είναι συναπόφαση, αλλά μοναδικά απόφαση του Κοινοβουλίου, διότι η συναπόφαση δεν θεμελιώνεται πουθενά εδώ. Άρα τι προσπαθούμε ε, να αναπτύξουμε μια τακτική προσέγγιση για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Το μόνο πράγμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε ως προνόμιο του Κοινοβουλίου στον καθορισμό της ίδιας του της έδρας ή των κανόνων οργάνωσής του είναι ότι προκύπτει από το γεγονός ότι εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς λαούς. Όπως γίνεται με όλα τα κοινοβούλια, ιστορικά, που εκπροσωπούν λαούς. Τα κοινοβούλια αυτά έχουν το δικαίωμα, το προνόμιο να καθορίζουν τους κανόνες τους. Είναι αυτή η λειτουργία της οργάνωσης. Οργανιζατσιόν σκεβάλτ στην γερμανική εκείνη θεωρία της κρατικής οργάνωσης και των κυρίαρχων κοινοβουλίων. Άρα εγώ δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε σαν να είναι θέμα συναπόφασης. Γιατί στο τέλος θα αναγνωριστεί ότι δεν είναι προνόμιο του Κοινοβουλίου. Και δεν θα μας εξυπηρετήσει. Αλλά καταλαβαίνω βέβαια το νόημα αυτής της τακτικής, της κινήσεως τακτικής. Έχω και τρίτο. Προσωπικό όμως. Είναι σημαντικό να μπει κάπου αυτή η ιστορική παραπομπή στην εξέλιξη των κοινοβουλίων και αυτό βάζω εγώ στην τροπολογία μου. Δηλαδή όλες οι βουλές από την Αγγλική Επανάσταση, από την Γαλλική Επανάσταση, όλα τα κοινοβούλια άλλαξαν τους συνταγματικούς κανόνες λόγω της άμεσης από μέρους τους εκπροσώπησης των λαών, βασισμένα σε αυτό δηλαδή. Αυτό ήταν πολύ σαφές μέσα στην εξέλιξη των συνταγματικών διαδικασιών και του Ενωμένου Βασιλείου στο 17ο αιώνα. Είναι πολύ σαφές αυτό. Το Κοινοβούλιο πήρε στα χέρια του τον καθορισμό των κανόνων. Το ίδιο και στα Ether Généraux, στην αρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Και αυτό διδάσκει και η ιστορία των βουλών μας απανταχού. Είναι μια εξουσία την οποία κατέκτησαν, δεν τους προσφέρθηκε μέσω συνθήκων, αλλά ήταν η δράση των μελών τους που εξασφάλισε την εξουσία αυτή. Τώρα βέβαια υπάρχει και η σχέση Κοινοβουλίου και Κομισιών μέσα στα, μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαισίου που πάντα προσπαθήσαμε να δώσουμε στο Κοινοβούλιο τον τρόπο, τη δυνατότητα να έχει έλεγχο των εκτελεστικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και είναι ενδιαφέρον ότι το Συμβούλιο, το οποίο επίσης εκπροσωπείται εδώ, είναι πάντοτε αντίθετο με αυτές τις συμφωνίες. Διότι αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ομαλή συνταγματική εξέλιξη. Βεβαίως με την εξαίρεση της ιστορικής περίοδου του Κρόμβελ, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν δεν πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, κανένας δεν θα αναγνωρίσει τις εξουσίες μας. Αν πιστεύουμε πραγματικά ότι εκπροσωπούμε, είμαστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να οργανώσουμε τα των εργασιών μας. Αν θεωρούμε πάντοτε ότι πρέπει να έχουμε σύμφωνες στις εθνικέ κυβερνήσει, τότε βεβαίως παρετούμεθα στην ουσία από την ιδέα αυτή της άμεσης εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σούλτ, μετά στον κύριο Μπράουντ. Και αφού κανεί άλλο δεν έχει ζητήσει το λόγο, θα ζητήσω από τον κύριο Χέφνερ να συνοψίσει. Α, και ο κύριο Ντάφ θέλει το λόγο. Ο κύριος Σάλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και δεν ήξερα ότι είχατε ξεκινήσει νωρίτερα τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ή τις τροπολογίες μας ε, τις θανάτωσε το αεροπλάνο. Ήμουν στο αεροπλάνο όταν έληξε η καταληκτική προθεσμία και γι' αυτό δεν πρόλαβα να τις υποβάλω. Εν πάση περιπτώσει θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για την σύνταξη αυτής της τόσο απαιτητικής έκθεσης. Ε, σε γενικές γραμμές και κατά κύριο λόγο συμφωνώ με την προσέγγιση σας. Οι τροπολογίες μου, εάν τις είχα υποβάλει, θα είχαν ως στόχο ε, όλα τα αριθμητικά στοιχεία, όλα τα νούμερα, όλα τα ερωτήματα να διαγραφούν υπό εάν αυτά θα οδηγούσαν ε, στην συναισθηματική εξέταση ε, του πράγματος. Εμάς μας απασχολεί το νομικό θέμα. Η Φλόγος είπε ότι είπε κάτι και είναι ε, μια προσωπική παρατήρηση αυτή ότι είναι ένα πολιτικό όργανο, ένα κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα να ε, αυτό οργανώνεται και να αυτό διατίθεται για το πού θα εδρεύει. Εμείς όμως δεν είμαστε ένα φυσιολογικό εντός εισαγωγικών κοινοβούλιο όπως τα εθνικά κοινοβούλια. Είμαστε κάτι πιο πρωτότυπο, ένα κοινοβούλιο sui generis στη δομή του και αντικατοπτρίζουμε ε, την τρέχουσα κατάσταση και τις ε, υφιστάμενες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το πώς και το πού θα οργανώσουμε ε, τη δουλειά μας είναι κάτι που θα πρέπει να ε, αποφασιστεί εμπλέκοντας όλους τους πολίτες και στις 28 πλέον χώρες ε, μέλη οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στη συζήτηση. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμβάλλουν ε, σε αυτή τη συζήτηση γνωρίζοντας με τι ακριβώ έχουμε να κάνουμε, αλλά και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και λοιποί. Όλοι γνωρίζετε και μάλιστα αναφέρεται και στην έκθεση το γεγονό ότι χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών. Ε, θα πρέπει να αλλάξει δηλαδή το πρωτογενές δίκαιο. Ιδαλλιώ δεν θα μπορέσουμε καν να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της αυτοδιάθεσης Και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα, ότι δηλαδή αυτή η έκθεση είναι μια συνεισφορά στην επικείμενη και πολύ αναγκαία ε, αλλαγή στη συνθήκη. Είναι μια συνεισφορά στη συζήτηση αυτή ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση και με τους πολίτες των κρατών μελών. Ιδαλλιώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε την ευκαιρία να την αλλάξουμε τη συνθήκη. Και υπό αυτή την έννοια επίσης συμφωνώ ε, με το εξή σημείο της έκθεσης που είναι και πολύ ενδιαφέρον. Το σημείο όπου ο κύριος Χέφνερ και ο κύριος Φόξ αναφέρονται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει την έδρα του και δεν παρεμβαίνει στον καθορισμό της έδρας των άλλων θεσμικών οργάνων, οι οποίοι, τα οποία ενδεχομένω έχουν την, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία και το δικαίωμα να ε, προβούν σε κάτι ανάλογο. Επομένως, πέρα από τη γραπτή και προφορική διαδικασία των τροπολογιών και των συμβαστικών τροπολογιών και του καθεξής, εμείς προσδοκούμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και να βρούμε συμβιβασμούς που θα οδηγήσουν τη συζήτηση στην κατεύθυνση που επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόντς, μετά στην κυρία Κιγιόμ, στον κύριο Σόφρον, μετά μια δεύτερη προσπάθεια από τον κύριο Νταφ, η κυρία Μπούζης και στο τέλος ο κύριος Χέφνερ, αλλά και ο Πλέγκοβιτς. Κύριε Μπρόντς, παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Ζήτω συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήμουν κι εγώ σε άλλη επιτροπή. Σίγουρα δεν μπορούσατε να παρηγορηθείτε με τίποτα λόγω της απουσίας μου. Εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να ταξιδεύει σαν τρελό, αν αυτό είναι που επιθυμεί, αλλά εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει την εξουσία να πάρει μία απόφαση οριστική, μια και καλή για το που θα εδρεύει. Είναι μια απόφαση που δεν επηρεάζει τα άλλα θεσμικά όργανα, επηρεάζει μόνο το ίδιο το Κοινοβούλιο και φυσικά και το φορολογούμενο ο οποίο εκπροσωπείται σε αυτό το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα άλλα θεσμικά όργανα να παίρνουν αυτή την απόφαση, ούτε καν να την παίρνουν από κοινού με εμάς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να διαλέξει που θα συνεδριάσει και θεωρώ και διορθώστε με αν ότι και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί επίσης να διαλέξει που θα συνεδριάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, που θα επιβάλλει στο Κοινοβούλιο να μοιραστεί και να λάβει από κοινού την απόφαση αυτή με άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, πολύ καλά. Κυρία Γκυγιόν, παρακαλώ για το θέμα αυτό. Ναι, και εγώ από τα μέλη που ήμουν ταυτόχρονα με στην Επιτροπή Δημοσιολευθεριών, καταλαβαίνετε, ζητώ συγγνώμη. Ναι, για την έδρα δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Αρκετές φορές εκφράστηκα και εδώ στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Διάβασα την έκθεση και διάφορες τροπολογίες και δεν ε, συμμερίζονται αρκετοί συνάδελφοι, κυρίως Γάλλοι, τις απόψεις αυτές αυτά που αναφέρονται ε, είναι και αφισβητήσιμα και λανθασμένα όπως θεωρούνται από ορισμένου ε, κυρίως για ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες όλα τα θεσμικά όργανα και για τον διαθεσμικό διάλογο, για τις συνθήκες ή τη διάφορα δια... στα... στοιχεία, τα στατιστικά, αναφερθήκαμε σε αυτά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες ομάδες, δεν μπορώ να πω την αποψή σας, αλλά για διάφορα θέματα, ε, τροπολογίες για το χρονοδιάγραμμα και άλλα θέματα. Θα δούμε κατά τις τροπολογίες τι θα γίνει. Ε, δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και σε κάποιους συμβιβασμούς, κάτι που δεν ε, χαράστε σαν προοπτική προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος. Thank you, Ακολουθώ τον κύριο Σόλτς, που ένα πράγμα σωστό που είπε είναι και στα πλαίσια της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολιτών. Αλλαγή των συνθήκων, αν γίνεται χάρη των πολιτών, που πάντως σε μένα βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο, τότε αυτή η έκθεση εκεί εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια ταυτόχρονα, θα δούμε και κάποια αντίσταση και από εθνικές βουλές και από μια τουλάχιστον χώρα μέλος. Άρα θα είναι πολιτική πραγματικά σύγκρουση. Καλά, έτσι είναι. Αλλαγή συνθήκης όμως σημαίνει επίσης ότι μπαίνουν στην ατζέντα και άλλα πράγματα. Και για αυτό το λόγο θα υπάρξει αντίσταση. Εγώ θεωρώ την αντίσταση εσφαλμένη. Πάλι αυτό είναι άλλη υπόθεση όμως. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι λάθος να διευρυνθεί η ατζέντα, να γίνει αλλαγή των συνθήκων και για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα που ενδεχομένως να προκύψουν και διότι η συνθήκη έχει αλλάξει με διάφορους τρόπους από την προηγούμενη συνέλευση. Και νομίζω συνέλευση είναι μια σωστή τομή διάδρασης μεταξύ Ένωσης και πολιτών. Και αυτό το είναι ένα σημαντικό στοιχείο για οποιαδήποτε αλλαγή συνθήκης ή άλλες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Συνέλευση πιθανόν να γίνει, όποιες και αν είναι οι αντιστάσεις, ίσως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κυρία Μπούσιτς, μετά ο κύριος Μπρένκοβιτς, μετά ο κύριος Νταφ και μετά ο κύριος Χέφνερ. Άλλος κανείς? Όχι. Ωραία. Εσείς. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ όλες και όλους. Είμαι νέο μέλος από την Κροατία και εγώ νομίζω βέβαια καταλαβαίνουμε τα αγγλικά Ήλπιζα ωστόσο να έχουμε και εδώ κροατική διερμηνία. Παρόλο που βεβαίω όλες και όλοι μιλούμε τις γλώσσες εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με όλο τον σεβασμό για τα όσα είπατε κύριε Πρόεδρε και επαναλαμβάνω ότι είμαι νέο μέλος, διάβασα ωστόσο το έγγραφο προσεκτικά και για τα όσα είπατε προηγουμένως, επαναλαμβάνω με όλο το σεβασμό που οφείλω στο αξίωμά σα, η θέση, η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ μπαίνει ένα θέμα συμβολισμού. Όλοι ξέρουμε την ιστορία και νομίζω ότι είναι σημαντικό το τμήμα αυτό της ιστορίας να μην λησμονείται και να λαμβάνεται υπόψη. Και ο συμβολισμός προκύπτει από αυτό. Δηλαδή, εκεί όπου συναντήθηκαν άνθρωποι που είχαν χωριστεί πριν από βαθιές διαφορές. Εγώ είμαι κροατισα και κατανοώ τη σημασία αυτής της προσέγγισης και τι σημαίνει να έχει κανείς ένα μέρος όπου να συνέρχεται μαζί με άλλους πρώην αντιθέτους. Δεν είναι και ασήμαντο αυτό που λέει η συμφωνία. και αυτά που λέτε εσείς βέβαια στο σχέδιό σας είναι σημαντικά. επαναλαμβάνω με όλο το σεβασμό που έχω για το όσα έχετε γράψει, νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Ορίστε. από την επόμενη συνεδρίαση τα κροατικά θα είναι γλώσσα εργασίας της παρούσης Επιτροπής. Εσείς κύριε Πρένκοβιτς. Συμφωνώ με την κυρία για την γλώσσα. Αφού είναι και συνταγματική επιτροπή εδώ, που αλλού να επιμείνει κανείς για να διαθέτει την 24η γλώσσα της Ένωσης. Μιας και είμαστε νέο εισερχόμενοι σε αυτή τη συζήτηση που κρατάει καιρό για την ενιαία έδρα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα μείγμα προβληματισμών που έχουν και σχέση με το οικονομικό και σχέση με την ε, εμφάνιση, με την εικόνα του Κοινοβουλίου και βεβαίως και με τις πρακτικές συνθήκες εργασίας των όσων εργάζονται στο Κοινοβούλιο με την έννοια ότι τόπος ε, λειτουργίας είναι και οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Επίσης το γεγονό ότι το Στρασβούργο δεν επιλέχθηκε κατά τύχη ενέχει κάποιο συμβολισμό και ιδίω σε μια χώρα εμείς μάλλον προερχόμενοι από μια χώρα η οποία υπέστη την επιθετικότητα άλλων στη δεκαετία του 90 και γνωρίζει τι θα πει συμφιλίωση. Έτσι λοιπόν εμείς βαθίζουμε προσεκτικά στη συζήτηση αυτή σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του θέματος και αν θα χρειαστεί τώρα τροποποίηση του πρωτο, πρωτογενούς δικαίου με κάποιο τρόπο τέλο πάντων είτε με τη διατύπωση που προτείνετε εσείς ή με διατυπώσεις που έβαλαν άλλοι στις τροπολογίες τους επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συνδέω λίγο την συζήτηση αυτή και με τη σχετικά πρόσφατη συζήτηση στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας για τις έδρες, δηλαδή 750 σημεία. Τώρα έχουμε φτάσει στις 766 έδρες στο Κοινοβούλιο. Απόφαση όμως που λήφθηκε πριν ενταχθούμε εμείς και επηρεάζει ορισμένους δικούς μας ευρωβουλευτές. Κάτι το οποίο δεν μας έχει ενθουσιάσει, να το πω έτσι απλά. Όπως είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε το πέρα δόθε, δύσκολο είναι και για μας να δικαιολογήσουμε το πώς μόλις μπήκαμε χάσαμε κιόλας έναν ευρωβουλευτή. Είναι, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα κύριε Τάφη, σας βεβαιώνω. διότι δεν είναι ευθύνη δική μας που μπήκαμε τόσο αργά με αυτή τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν είχαμε το πλήρη αριθμό των ευρωβουλευτών που προβλεπόταν αρχικά θα ήταν πολύ διαφορετική και η στο κροατικό κοινό. Όλα αυτά τα λέω τέλος πάντων διότι θέλω να πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη περίσκεψη. Να δώσω στον κύριο Νταφ ε, μια δεύτερη ευκαιρία. Παρακαλώ. Να διευκρινίσω κάτι που είπε ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει πού θα συνεδριάσει το ίδιο. Αυτό έχει θεσπιστεί στο πρωτόκολλο υπαριθμών 6, ότι θα συνεδριάσει διάφορα μέρη κτλ. και βεβαίως τα κράτη-μέλη είναι οι άρχοντες των συνθήκων. Και ακριβώς αυτό επιθυμώ εγώ να αλλάξει. Με συγκλώνησε όταν διάβασα για το 17ο αιώνα στην Αγγλία και για την κοινοβουλευτική παράδοση τότε τότε ήταν καιρή επαναστατική. Πολεμούσαμε εναντίον της ε, ολιγαρχίας. Και αυτό το οποίο έπρεπε το Κοινοβούλιο να καταφέρει είναι να εδρεώσει το δικαίωμα αυτό να συνέρχεται, να συνεδριάζει, να ε, συγκεντρώνονται τα μέλη, να συναθρίζονται και δεν τους διέφερε καθόλου το που ήθελαν μόνο να μπορέσουν να ε, συνεδριάσουν σε κάποιο μέρος ασφαλές και σχετικά κοντά στην αυλή. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η ε, γυτνίαση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στην περίπτωση αυτή. Καλό είναι τα σημαντικά μαθήματα του, της ιστορίας του 17ου αιώνα να τα ισορροπούμε, να τα φέρνουμε σε ένα σημείο ισορροπίας με τις ε, πολύ σημαντικές συνέπειες που είχε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του 20ου αιώνα, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να τροποποιηθεί, να εξυγχρονιστεί για να εξυγχρονιστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να καταστεί και περισσότερο αποτελεσματικό. Δεν πιστεύω ότι το γεγονός ότι υποχρεωνόμαστε να συνεδριάζουμε στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή είναι συνταγματικό σκάνδαλο ή πλήγμα όνειδος για τη δημοκρατία, πιστεύω πολύ απλά ότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα αυτό και μόνο. Είναι κουραστικό και μας απομακρύνει ακόμα περισσότερο από εκεί όπου εδρεύει η εξουσία. Και θα ήθελα οι Γάλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι πολύ ορθώς μάλιστα, και σαφέστατα υπερασπίζονται το Στρασβούργο ως έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουν και εκείνοι με τη σειρά τους όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, και δεν νομίζω ότι το έχουν πράξει αυτό ακόμα. Ε, έχουν συμπεριλάβει δηλαδή την εξέταση αυτών των ζητημάτων στην επιχειρηματολογία που προβάλλουν. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, πολύ ωραία. Είχαμε μια πολύ ολοκληρωμένη συζήτηση. Όλοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Κύριε Χέφνερ, μπορείτε να συνεψίσετε από πλευράς ε, των ε, συνεισηγητών, ημών και ημών. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ για την πλούσια και διαφοροποιημένη συζήτηση. Ιδίως ευχαριστώ τον κύριο Δρούτσα, Νταφ, Ραμζέλ, Σόλτς, τον κύριο Μπρόνς, τον κύριο Γκιόμ, Σέφλιν, Μπούσιτς και τον κύριο Μπρένκοβιτς. Ε, χαίρο άλλωστε που ήρθατε και στο μέλλον να συνεργαστούμε. Καλώς λοιπόν. Μία παρατήρηση αν με επιτρέπετε. Αναφέρεται στα λόγια των δύο Κροατών συναδέλφων που τονίσατε με ιδιαίτερη έμφαση την ιστορία της Ευρώπης που κατέληξε στην απόφαση που γνωρίζουμε καθώς και την αξία να διδασκόμαστε από την ιστορία. Είναι σημαντική αυτή η υπόδειξη. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι, από τα διδάγματα, όχι, ότι στα διδάγματα της ιστορίας μάλλον εντάσσεται και το δίδαγμα να αγωνιζόμαστε διαρκώς υπέρ της δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο τούτο, εδώ το κοινοβούλιο αν τη δική του ιστορία, έχει αγωνιστεί και εξακολουθεί και αγωνίζεται. Αυτό δεν ήταν έτσι από την αρχή. Από την αρχή ήταν μοναχά διακυβερνητική συνεργασία. Κάποια στιγμή μπήκε στη μέση το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο αποφάσισε πού θα διαθέτει την έδρα του. Τότε υπήρχε ακόμη, όχι Κοινοβούλιο, αλλά μια μη εκλεγόμενη συνέλευση, καμιά εξινταριά μελών, συγγνώμη, περίπου, που δεν είχε απολύτω καμία αρμοδιότητα το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε και κατέκτησε δικαιώματα, το δικαίωμα να εκπροσωπεί τους λαούς με τις άμεσες εκλογές κτλ. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι όχι μόνο νομιμοποιούμενη η διαφωνία αυτή, αλλά και απαραίτητη. Δηλαδή, με την νέα αυτή κατανόηση του ρόλου του Κοινοβουλίου ως ισότιμου συνομοθέτη με το Συμβούλιο. Δεν είναι ορθό ότι το Κοινοβούλιο επιλέγει όχι μόνο την έδρα του, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του. Και επομένως, επομένως της αυτοοργάνωσης του. Ο Άντριου Νταφ μίλησε για το Συμβούλιο. Ναι, για το Συμβούλιο υπάρχει ρύθμιση του πρωτοκόλλου υπαρθμών 6. Το Συμβούλιο όμως τηρεί πολύ λιγότερο τα προβλεπόμενα του το πρωτόκολλο 6 από ό,τι το κοινοβούλιο. Βεβαίω μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει προσφυγέ. Για μα, ωστόσο, έγινε προσφυγή για το χρονοδιάγραμμα του κοινοβουλίου. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε αν δεν σας αρέσει όπως είναι, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνθήκες. Μέσα στα πλαίσια των υφισταμένων συνθήκων δεν υπάρχει τρόπος άλλος, είπε το δικαστήριο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητούμε τώρα. Κοιτάξτε, τώρα ευχαριστώ και για τις τροπολογίες που βάλατε και οι οποίες δεν παρουσιάστηκαν όλες. 124 συνολικά τον αριθμό, 92 από Γάλλους Ευρωβουλευτές, 32 από όλες τις υπόλοιπες 27 χώρες εδώ μπορεί να δώσει κανείς διαφορετικές ερμηνείες. Μπορεί να πει κανείς ότι όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ συμφωνούν. Μπορεί να πει κανείς ότι θίγονται διαφορετικά οι μεν και οι δε. Εδώ έχω μια παρατήρηση να κάνω. Εμείς δεν κάναμε έκθεση, ούτε θα κάνουμε μια έκθεση προς Θεού υπέρ ή κατά μιας χώρας. Εμείς κάνουμε μια έκθεση, φτιάχνουμε μια έκθεση που απευθύνεται σε όλους τους ευρωβουλευτές και τους επηρεάζει όλους. Η ρύθμιση που έχουμε τώρα μας επηρεάζει όλους και όλες. Με διαφορετικό τρόπο βεβαίω. Και οποιαδήποτε αλλαγή πάλι θα μας επηρεάσει όλους. Γι' αυτό νομίζω τέτοιες αλλαγές οφείλουμε να τις συζητήσουμε ήρεμα, νυφάλια και δημοκρατικά. Ωστόσο προσοχή. Στην συζήτηση περί της έκθεσης αυτής να μην πιάσουμε τα εθνικά χαρακόμματα δεν τίθεται θέμα εθνικότητας, αλλά κατανόησης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ερωτήματος της συνταγματικής του θέσης, καθώς επίσης και των επιπτώσεων για τις φυστάμενες ρυθμίσεις και απέναντι στην ιστορία, αλλά και για θυγόμενες χώρες, περιφέρειες και Το Κοινοβούλιο πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να τα συζητήσει τα πράγματα αυτά με τρόπο αξιοπρεπή και που να Έρετε στο ύψος των περιστάσεων. Έχω σημειώσει τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι και για λόγους χρόνου δεν θα απαντήσω σε όλες και όλους ξεχωριστά. Θα κάνω καλύτερα κάτι άλλο. Θα εξηγήσω με λίγα λόγια το περιεχόμενο των τροπολογιών, που για μας είναι σημαντικές. μία ομάδα τροπολογιών, η 3, 24, 46, 94, 97 και 105 και άλλες, που αναφέρονται στο θέμα του πολυκεντρισμού. Με την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σε ένα τόπο ή σε διαφόρους τόπους. Τέθηκε εκεί το θέμα και των εδρών άλλων οργάνων. Οι συνεισηγητές αποφασίσαμε τον προβληματισμό των εδρών άλλων οργανισμών να τον αφήσουμε απ' έξω. Και δεν θελήσαμε να πούμε τίποτε καθαρά για οποιοδήποτε άλλο όργανο. Διότι αφενός θεωρούμε ότι δεν νομιμοποιούμεθα και επίσης διότι δεν θέλουμε να τα εξισώσουμε όλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μοναδικός οργανισμός, το μοναδικό όργανο το οποίο εκλέγεται ευθέως από όλους τους πολίτες της Ένωσης και επομένω οφείλει να τύχει και άλλη μεταχείριση από τα άλλα όργανα. Και το ζήτημα αυτό του πολυκεντρισμού είναι δικαιολογημένο. Εγώ κατανοώ πολύ καλά την θέση των προσώπων που λέγουν αυτά και πρέπει να ενταχθεί μέσα σε μια δημοκρατική διαδικασία αναζήτησης διαμόρφωσης άποψης. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί καταλήξει τελικά να ρυθμίζει τα του οίκου του, πρέπει να βρεθούν λύσεις και για τα άλλα. Αυτό είναι δημοκρατικό. Έσως να υπάρξει μια πολύ κεντρική ρύθμιση λοιπόν εν τέλει. Υπάρχει και ένας αριθμός τροπολογιών που αναφέρεται στις υπογραφές είναι 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 74 μέχρι 78 και 82. Πολλές από αυτές λένε ότι ε, η σχετική αναφορά για, με τη συλλογή υπογραφών κτλ δεν είναι αναφορά ή πάντως δεν είναι παραδεκτή. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό στην παρούσα Επιτροπή, διότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας. Προτιμώ την υπόθεση αυτή να τη συζητήσει η Επιτροπή Αναφορών. Ρωτήσαμε και γραπτά και προφορικά την γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών και η απάντηση που μας έδωσε είναι ότι έλαβε η Επιτροπή Αναφορών την αναφορά αυτή, ότι η γραμματεία την θεώρησε παραδεκτή, ότι συζητείται αλλά δεν έχει ακόμα κρυθεί η μοίρα της. Είναι ακόμη ανοιχτή. Εμείς αναφερόμεθα στην διαδικασία, είναι σημαντικό αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο να κρίνουμε δραστηριότητες πολιτών. Τώρα, υπάρχουν και πολλές τροπολογίες που αναφέρονται στο κόστος. 6, 7, 8, 15, 53 μέχρι 70, 81, 93, 112 και μέχρι 124 κτλ. Εκεί έχουμε το πρόβλημα που είπε ο Άσλι Φόξ στην αρχή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πραγματικά νούμερα τα οποία να είναι αντικειμενικά βέβαια, αντικειμενικά βεβαιωμένα και σίγουρα ορθά για το κόστος των δύο εδρών σε σύγκριση ή και τριών μάλιστα σε σύγκριση σε αντιπαραβολή με μια έδρα. Ρωτήσαμε παντού, το πρόβλημα είναι ότι δεν λάβαμε καμία συνολική πραγματικά θεμελιωμένη απάντηση. Βεβαίως με τα νούμερα μπορεί κανείς να αποδείξει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένας αριθμός 51 εκατομμύρια που προέρχεται από την διοίκηση του Κοινοβουλίου. Βέβαια, ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει πολλά στοιχεία κόστους τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει και το κόστος της συντήρησης των κτίριων... που μένουν 320 μέρες τον χρόνο κενά, ούτε το κόστος για τον τεχνικό εξοπλισμό, κομπιούτερ κλπ ούτε το κόστος για τη μετακίνηση των πολιτικών ομάδων, ούτε των δημοσιογράφων και άλλων εκπροσώπων των ε, μέσων ενημέρωσης που σε μεγάλο αριθμό και βαθμό πληρώνονται από το ίδιο το Κοινοβούλιο και επομένως θα προκύψουν αλλαγές εκεί. Το πρόβλημα για μας είναι ότι πάλι από το ίδιο το Κοινοβούλιο, από την Joint Working Group που αποτελείται από Προεδρείο και Επιτροπή Προϋπολογισμών, το 2012 προέκυψε ένα ποσό 148 εκατομμυρίων που αναφέρεται υποτίθεται στα πριν από την προς Ανατολάς διεύρυνση της Ένωσης και που θα αυξάνονταν συνολικά υποτίθεται με την ένταξη των ανατολικών χωρών. Α, μια στιγμή σε 169 εκατομμύρια μια στιγμή να ελέγξω ε, νομίζω ότι δεν έχω το σωστό έγγραφο μπροστά μου σας τα έχω βάλει σε ένα ξεχωριστό σημείωμα τα 169 εκατομμύρια ήταν για το έτος 2002 όπου ακόμα δεν συμπεριλάμβαναν το κόστος της προσανατολάς διεύθυνσης. Και βεβαίως μετά την ε, διεύρυνση προσανατολάς... θα ανέρχονταν σε ένα των 200 εκατομμυρίων. Τι να κάνουν στην περίπτωση αυτή οι συνεισηγητές. Βάλαμε αυτό το πλαίσιο που προκύπτει από τα νούμερα που λάβαμε από Προεδρείο και Επιτροπή Προεπολογισμών. Η επιθυμία που έχουμε εμείς είναι να υπάρξουν επιτέλους οι σχετικοί αριθμοί σε ένα έγγραφο που να προκύπτουν από μια μεθοδολογία υπολογισμού που να μην εμφισβητείται από κανένα. Αυτά για το κόστος. Συντομεύω λίγο. Υπάρχει και ένας αριθμός τροπολογιών για την τροποποίηση των συνθήκων, αν δηλαδή μπορούμε να προτείνουμε τροποποίηση των συνθήκων, είναι οι τροπολογίες 99, 100, 101 και μέχρι 119. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να τον βαδίσουμε όμως ευθέως. Εγκρίθηκε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού και όχι σύμφωνα με το άρθρο 74. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Άνδριο Ντάφ πριν, διότι βεβαίως μια διατύπωση σαφέστερη θα ήταν προς όφελος και των συνεισηγητών. Θα δούμε, ίσως την περιλάβουμε και σε μια προσπάθεια συνενετικών τροπολογιών, συμβιβαστικών τροπολογιών δηλαδή. Βεβαίω το ερώτημα που τίθεται είναι ποια θα είναι η νέα διαδικασία. Το Κοινοβούλιο θα λάβει το δικαίωμα να αποφασίζει μόνο του, όπω είπε ο Παύλο Ραουζελ και άλλοι, είναι ζήτημα αυτοοργάνωση, δικαιώματο αυτοδιαχείρισης μέσα σε μια δημοκρατία και απορρέει από το άρθρο 10 της συνθήκης για παράδειγμα ή θα πρέπει να είναι κάποια διαφορετική διαδικασία λήψης αποφάσεως, όπως για παράδειγμα μια συνενετική διαδικασία. Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από διάφορες παραλλαγέ. Όσον αφορά όμως ποια είναι η πρόταση που θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο, οι συνεισηγητέ τονίζουμε ότι το Κοινοβούλιο στην συζήτηση αυτή θα πρέπει να προχωρήσει με την αξίωση να λάβει το ίδιο το δικαίωμα να αποφασίζει. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό η συζήτηση αυτή να γίνει με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από την παρούσα κατάσταση όπου εάν δεν καταλήξουμε σε ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Θα πρέπει να είναι ένας δρόμος που να μπορούμε να τον πατήσουμε όχι μόνο νομικά αλλά και στην πράξη και το Κοινοβούλιο και στην θέση που είχε εκφράσει πριν από την τελευταία συνέρευση δηλαδή να αποφασίζει μόνο του για τα πράγματα αυτά, αυτή νομίζω θα πρέπει να είναι η θέση υπέρ της οποίας θα πρέπει να ταχθούμε και εμείς ως Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ως Κοινοβούλιο. Θα πρέπει βεβαίως αυτή η θέση να γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας διακυβερνητικής συνέλευσης. Και βεβαίως είναι δυνατό ή οδήποτε αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών να προσεγγίζει πολύ σε αυτά που ορίζει ο Άντζιου Νταφ σήμερα ως απέτηση του Κοινοβουλίου. Δεν σας εξήγησα όλες τις τροπολογίες. Για λόγους χρόνου αρκούμε σε αυτά. Ο Άσλι Φόξ και εγώ θα εξετάσουμε πραγματικά σε βάθος όλες τις τροπολογίες σας και στη διάρκεια των θερινών διακοπών θα καθίσουμε να δούμε πού μπορούμε να βρούμε συμβιβασμούς. Και μετά από μια νέα συζήτηση το φθινόπωρο θα καταθέσουμε συμβαστικές τροπολογίες για να ψηφιστούν. Μία τελευταία σκέψη, αν με επιτρέπετε, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδίως εμείς ως Συνταγματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο να διεξάγουμε τη συζήτηση με έναν τρόπο, αλλά και να αναζητήσουμε έναν τρόπο που δεν θα μας αποδυναμώσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα μας διασπάσει στα, στις διάφορες γραμμές διάσπασης που δεν είναι μοναχα η εθνική, αλλά να το συζητήσουμε με έναν τρόπο που εν τέλει να μας ενώσει στα πλαίσια μιας αξίωσης που θα προβάλλει το Κοινοβούλιο στη συζήτηση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Έτσι ώστε μέσα στην προσπάθεια διαρκούς καλλιέργειας και εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να καθορίζει και την έδρα του και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του. Αυτό θεωρώ ότι είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι είναι και πρωτίστως η επιθυμία που εφράζουν οι πολίτες μας απέναντι σε εμά. Στην τελευταία εκλογή θα έλεγα σε κάθε δεύτερη δημόσια συνάντηση που συμμετείχα, μου τίθεται το, ερώτημα γιατί ταξιδεύετε διαρκώς μεταξύ Βελγίου και Στρασβούργου, Βρυξελών και Στρασβούργου. Δεν το κατανοούν οι πολίτες. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως απορριπταίο και λόγω του κόστους και για διάφορους άλλους λόγους. Και όταν εξήγησα ότι τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λέτε αλλά το Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει, τότε κούνησαν με απορία τα κεφάλια τους και είπαν «Μα τι κοινοβούλιο είναι αυτό» που δεν μπορεί καν αυτό να αποφασίσει. Αν όμως το κοινοβούλιο δεν πει ότι στο μέλλον θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε, τότε και στις επόμενες ευρωεκλογέ θα έχω μέγιστες δυσχέρειες να εμφανιστώ ενώπιον των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να αναμετρηθεί με τα θέματα αυτά, να διεξαγάγει τη συζήτηση και να φέρει την συζήτηση αυτή σε ένα πέρας και όχι να παρατείνει πράγματα επί δεκαετίες τα οποία στην πράξη δεν αντέχουν πλέον και βεβαίως δεν γίνονται διόλου κατανοητά από τους πολίτες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Κέρχαλτ. Τα μέλη πρέπει να γνωρίσουν ότι Μέχρι τις 19 Ιουλίου όλες οι τροπολογίες θα είναι μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες. Θα συζητήσουμε ε, τις συμβιβαστικέ τροπολογίες στις 17 Σεπτεμβρίου, θα ψηφίσουμε στις 14 Οκτωβρίου και ελπίζουμε ε, να πάει το θέμα στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Τώρα, η Παολίνα εν ώψη της 17ης Σεπτεμβρίου θα έρθει σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές για να κανονίσει τις συνεδριάσεις. Έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση, διότι το σημείο 6 έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ.